όργανο στην Πορτογαλία κάνει ό,τι μπορεί σε συνεργασία με την ΕΟΚΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εν τέλει θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών, μια Ευρώπη των περιφερειών. Χαίρομαι που κατορθώσαμε να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση όσον αφορά την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Μάλιστα, καταφέραμε να καταργήσουμε τις συγκρούσει συμφερόντων μεταξύ αυτού του μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων. Μπορούμε να φτάσουμε σε εγγύσεις έως και 100% σε σύγκριση με το 75% της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο συνεισηγητή, ο κύριος Γκουαλτιέρη, ο οποίος απουσιάζει όμως. επομένω, δίνω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Μπιενκόφσχα. Αξιότιμα μέλη, η σημερινή συζήτηση για το πρόγραμμα Invest EU στην ε, τελευταία αυτή ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια βληματική συζήτηση για την υποστήριξη που δίνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των επενδύσεων. Εξ ονόματο λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Η μερική συμφωνία, στην οποία καταλήξατε πολύ γρήγορα με το Συμβούλιο για το Invest EU, θα επιτρέψει την γρήγορη προπαρασκευαστική εργασία Κατά αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος αυτού στο πλαίσιο του επερχόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το πρόγραμμα InvestEU πρόκειται να απλουστεύσει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και με μια ενιαία εγγύηση, με ένα ε, ενιαίο σύνολο κανόνων θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να καλύψουμε επενδυτικά κενά και να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Θέσεις απασχόλησης, ενεργειακή απόδοση, αστικές μεταφορές είναι ορισμένοι από τους τομείς ε, για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις. Η εγγύηση για το πρόγραμμα Invested Youth θα επιτρέψει τις επενδύσεις αυτές και θα κινητοποιήσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για το δημόσιο καλό. Το Ταμείο αυτό θα υποστηριχθεί από το συμβουλευτικό όργανο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμώ επίση το γεγονό ότι οι συνομοθέτε υποστήριξαν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρχει μια εγγύηση από τον ενωσιακό προπολογισμό. Ο στρατηγικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πλέον ε, έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο του κανονισμού και να γνωρίζετε καλύτερα η εμπειρογνωμοσύνη τη τράπεζα αυτή, αλλά υπάρχουν πλέον και άλλοι παράγοντε όπω διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπω ε, η EBRD, η ε, Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι εθνικές επενδυτικές προθετικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν εταίροι υλοποίηση. Κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε όλη τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη με έναν τρόπο συμπληρωματικό, συνδυαστικό, προκειμένου να έχουμε καλύτερη γεωγραφική κάλυψη και να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η προετοιμασία του προγράμματος αυτού αλλά και η εφαρμογή του θα φέρει κοντά τους παράγοντες αυτούς θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν την κυριότητα του συστήματος αυτού και να διαμορφώσουν το μελλοντικό πρόγραμμα Invest in You. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε Μακροπρόθεσμου ισχυρού επενδυτέ οι οποίοι θα υποστηρίσουν του βασικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη πολιτική καθοδήγηση στο πρόγραμμα InvestEU, η απαραίτητη λογοδεσία, η απαραίτητη διαφάνεια και προκειμένου να αυξηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Θεωρούμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα αυτά τα σημεία βελτιώνουν την νομοθετική πρόταση. Πρέπει να πω ότι ε, εκτιμούμε πάρα πολύ τι σημαντικότερε προσπάθειε που κατέβαλαν οι δύο συνεισηγητέ, οι σκιώδει εισηγητέ και οι δύο εμπλεκόμενε επιτροπέ, προκειμένου να καταφέρουμε πάρα πολύ γρήγορα σε ένα πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Δράτω με τι ευκαιρίε προκειμένου να ευχαριστήσω και τη Ρουμανική Προεδρία για τι προσπάθειε που κατέβαλα και αυτή. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης, που είναι η κυρία Τζεντίλε. Αλλά από ό,τι βλέπω, έρχεται ο συνεισηγητής. Ίσως θα σας δώσω λοιπόν το λόγο μετά, κυρία Τζεντίλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δίνουμε τη δυνατότητα στους ε, Ευρωπαίους πολίτες να δούνε ξεκάθαρα ότι αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε, συχνά, περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο από μια πολιτική λιτότητος προς μια πολιτική επενδύσεων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, όλο και περισσότερο στρεφόμαστε προς την βιωσιμότητα, προς την ε, αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω του προγράμματος Invest in You μπορούμε να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, μπορούμε να προωθήσουμε φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές ή την κυκλική οικονομία. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε σχολεία, πανεπιστήμια, καταρτήσεις ε, για νέες θέσεις απασχόλησης. Μπορούμε να ενισχύσουμε επίσης τη δημόσια υγεία, την υγειονομική περίθαλψη. Μπορούμε να προωθήσουμε την κοινωνική οικονομία και να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Το πρόγραμμα InvestEU είναι ένα πρόγραμμα υπέρ των πολιτών και λαμβάνει υπόψη πραγματικά την ευημερία και την καλή διαβίωση όλων των πολιτών σε όλες τις πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ένα πρόγραμμα το οποίο βάλει κατά της φτώχειας. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη, το συνεισηγητή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματική χαρά για μένα να μπορώ να παρουσιάζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πόρισμα μιας ε, άοκνης ε, προσπάθειας που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες και που έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου, Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε, καθώς επίσης και όλους τους και οδησηγητές και όλους όσοι συνέβαλαν προκειμένου το κείμενο αυτό να βελτιωθεί. Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε η οικονομική κρίση, είχαμε την πολιτική λιτότητος και κατά αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν πάρα πολύ οι δημόσιε αλλά και οι ιδιωτικέ επενδύσει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία πρωταρχική μα λοιπόν προτεραιότητα ήταν να δώσουμε νέα όθηση στι επενδύσει, περισσότερε επενδύσει ω βασική προπόθεση για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη χάρη σε μια ευέλικτη ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας και χάρη σε νέες πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων καταφέραμε να διορθώσουμε την ακολουθούμενη πολιτική οικονομίας. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πολλά επενδυτικά κενά όσον αφορά την καινοτομία, όσον αφορά τις υποδομές, υλικέ και άειλε ε, όσον αφορά τι κοινωνικέ πολιτικέ και όσον αφορά την πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Όλε αυτέ οι προκλήσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ και ελπίζουμε θα τι αντιμετωπίσουμε τώρα με το νέο αυτό πρόγραμμα InvestEU. Ενισχύουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στον τομέα τη έρευνα, στον τομέα τη καινοτομία, τις βιώσιμες υποδομές και θεωρούμε ότι με το πρόγραμμα αυτό, το InvestEU, θα καταφέρουμε να καλύψουμε τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις κοινωνικές υποδομές και θα καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε πολλά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής στέγασης. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Συμβούλιο επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, καταφέραμε να θεσπίσουμε ότι το κόστος της εγγύησης για τους ε, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνδέεται με το προφίλ του κινδύνου των συγκεκριμένων οικονομικών επενδύσεων και ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε επενδυτικές πλατφόρμες και να προωθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις στις περιοχές εκείνης Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα επενδυτικά κενά. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να επέμβουμε μέσω επενδύσεων στι περιοχέ εκείνε οι οποίε υπολείπονται σε σχέση με τι υπόλοιπε πιο προηγμένε περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι δίδεται μέσω τη νέα αυτή πρόταση ένα πιο κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και στι εθνικέ επενδυτικέ τράπεζε, προκειμένου να μπορούν και αυτέ να συμβάλλουν στο επενδυτικό αυτό πρόγραμμα. Οι εθνικέ αυτέ τράπεζε πρόθεση θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην ενωσιακή εγγύηση και κατά αυτόν τον τρόπο του δίδεται μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων που μπορούν να έχουν πολύ θετικέ επιπτώσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Τέλος, καταφέραμε να θεσπίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν όχι μόνο τη δυνατότητα να δίνουν μέρος των πόρων τους στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και κατ' επέκταση έπειτα στο πρόγραμμα Invest in You, αλλά θα μπορούν να συνεισφέρουν και με επιπρόσθετους πόρους που ε, κατά προτεραιότητα θα θεωρούνται κατά αποκοπήν ε, συνεισφορές στο πρόγραμμα και επομένω δεν θα συνυπολογίζονται στον ε, υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματος στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το κείμενο λοιπόν το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο κείμενο και απαιτείται αυτή τη στιγμή ένα 55% των επενδύσεων να συμβάλλουν στους στόχους που προβλέπονται στην Συμφωνία των Παρισίων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το απαραίτητο επενδυτικό θετικό κλίμα, να υπάρχει απαραίτητη προβλεψιμότητα όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό InvestEU να συνάδει περισσότερο με τη χρηματοδότηση η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι ισχυρή στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το πρόγραμμα Invest in You είναι ένα πρόγραμμα καθοριστικό, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί την μόνη πολιτική προτεραιότητα για την επόμενη α, κοινοβουλευτική θητεία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σφαιρικό επενδυτικό πρόγραμμα, προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική βιωσιμότητα, την απασχόληση και την καινοτομία. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο έχει εκ μέρους του ΕΛΚΑ ο κύριος Κάρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συγητές, Φερνάντες Γκουαλτιέρη. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους ε, ε, και να πω ότι και ο τον Μπούλμαν και εγώ ξεκινήσαμε μαζί με σας αυτόν τον αγώνα για τις επενδύσεις. Σίγουρα ε, δεν είναι ένας ε, αγώνας ε, ταχύτητας, αλλά ένας μαραθώνιος. Ξεκινήσαμε με το σχέδιο Juncker αυτό το μαραθώνιο, που ήταν η πρώτη πρωτοβουλία. Έπειτα είχαμε το FC2 που βελτίωσε τα πράγματα και έχει επιμηκυνθεί η ισχύ του μέχρι το 2020. Θέλουμε επίσης να δούμε και τι γίνεται με τις χώρες γειτονία και για την Αφρική. Και κλείνουμε τώρα αυτή την νομοθετική θητεία με ένα επόμενο κεφάλαιο μέχρι το το 2027 το InvestEU 200 ε, δις ε, ε, ευρώ επενδύσεων προωθήθηκαν 954.000 επιχειρήσεις μπορούν να υποστηριχθούν και μέχρι στιγμής έχουμε κινητοποιήσει 50 δις και θα έχουμε και πολύ περισσότερα ε, κέρδη. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Με το InvestEU Έχουμε ε, επίσης ε, έναν πολύ αποτελεσματικό στόχο, ε, τη μείωση της γραφειοκρατίας, συνοχωνεύοντας τα 14 αυτά εργαλεία σε ένα. Και επίσης ενισχύουμε και την εφαρμογή των στόχων για το κλίμα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε αυτό το 25% τουλάχιστον των εγγύσεων που θα πρέπει να συνεισφέρουν προς αυτό το στόχο. Επίσης βελτιώνουμε την παροχή συμβουλών, την υποστήριξη και αυτών που που συμμετέχουν σε σχέδια, σε έργα μικρής ε, κλίμακας και έχουμε επίσης την εγγύηση αυτή ε, που την επενδύουμε και σε μικρότερα Ινστιτούτα, ε, σε μικρότερα ιδρύματα. Επίσης βελτιώνεται η διαφάνεια των επενδυτικών αποφάσεων. Το InvestEU όμως δεν είναι το τέλος, είναι αν θέλετε το τέταρτο ορόσημο, είναι το τέταρτο στάδιο που θα ενισχύσει ε, τις επενδύσεις από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι και στην επόμενη ε, θητεία θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκλοανέκα Μωρά εκ μέρους Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά και εγώ θέλω να χαιρετήσω το έργο των συνεισηγητών. Η μερική προσωρινή αυτή συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU στο πλαίσιο βεβαίως του ΠΔΕΛΤΑΠΗ 2021-2027 είναι ένα ηχηρό θετικό μήνυμα που ε, είναι υπερήφανο που στέλνει προς ε, το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη και του, σε επιτυχία του πρώτου επενδυτικού προγράμματος του σχεδίου Juncker για πολλαπλασιασμό των επενδύσεων με δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βιώσιμη ανάπτυξη από τον Ιανουάριο του 2021. Έτσι η χρηματοδότηση για τοπικά έργα θα προωθηθεί τομέα της έρευνας, των βιώσιμων υποδομών, ψηφιοποίηση, στήριξης ΜΜΕ, κάτι πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως θεσπίζεται και η εγγύηση που βάζει και έναν ηθικό βιώσιμο χαρακτήρα στην επένδυση. Και αυτό είναι σημαντικό. Μιλάμε για σημαντικέ εταιρικέ σχέσεις μεταξύ ε, ΤΕΠΑ, ε, Κομισιών, και ε, εθνικών και τοπικών επενδυτικών τραπεζών για την πρώτη περιβαλλοντικών κοινωνικών έργων που επιλέγονται ε, για να σεβαστούμε τους στόχους των Παρισίων και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΠΑ. Μία παρατήρηση έχω ε, που αφορά το τέταρτο σκέλος για το οποίο έκανε λόγο ο κύριος Φερνάντες που λέει ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε κοινωνικές ε, επενδύσεις, επενδύσεις στις διάφορες αρμοδιότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους κλάδους των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να σχετιστούν με το θεματολόγιο τον πολιτισμό που δεν μπορεί να μείνει εκτός ε, του διαλόγου. Ε, πρέπει επίσης να στραφούμε ε, εμείς στους πολίτες, γιατί η Ευρώπη έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα απλό χρηματοδοτικό εργαλείο πρέπει να είναι φαλτήριο προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, ακολουθεί αυτές τις αλλαγές και θα οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή ε, παραδείγματος. Θα πρέπει επίσης να είμαστε προοδευτικοί είναι μια Ευρώπη που θέλουμε να δημιουργήσουμε που θα είναι κοντά στους πολίτες, δίνοντας συγκεκριμένες ελπίδες και φιλοδοξία. Ε, ε, ε, Πάκετ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, InvestEU. Θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία. Περίπου 40 δισεκατομμύρια με τη μορφή εγγυήσεων, δεν πρόκειται για επιχορηγήσεις. Πολλές επενδύσεις θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σε πολλούς τομείς οι ευρωπαϊκές εταιρείε θα τύχουν υποστήριξη και θα μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα. Δεν θα εξαρτώνται από εξωευρωπαίους δωρητές. Θα γίνει μια σύμπηξη λοιπόν των εφισταμένων χρηματοδοτικών επενδυτικών μηχανισμών. Αυτό είναι εξαιρετικό. Τα πάντα πλουστεύονται. Οι εθνικές προθερικές τράπεζες αποκτούν σημαίνοντα ρόλο. Οι φλεμαδικές τράπεζες θα έχουν σήμερα τον ρόλο και στη δική μου χώρα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα λοιπόν είναι έκτακτο, έξοχο. Η αλλαγή αυτή θα φέρει αποτελέσματα. Πρόκειται για την τελευταία μας ολομέλεια βεβαίω. και πιστεύω ότι τελειώνουμε πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της ομάδας Άλντε, κυρία Βίρινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε καταρχάς το ΕΦΣΙ και τώρα το InvestEU, το οποίο θα δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και στην επόμενη θητεία. Και δείχνει μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Ένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε από την κρίση του 2008 είναι ότι η σταθερή οικονομία συνιστά ε, μια οικονομία των επενδύσεων. 650 σε, σε παραπάνω επενδύσεις λόγω του προγράμματος. Και αυτό είναι μια υπόσχεση για το μέλλον. Ιδίω στην καινοτομία, στην έρευνα, στην ψηφιοποίηση. Έτσι, η Ένωσή μας την επόμενη ε, περίοδο, προγραμματική περίοδο, θα γίνει ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη στον κόσμο για τους επενδυτές, για τα δημιουργικά μυαλά και για το εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, ας δώσουμε ένα τέλος στο κενό αυτό που υπάρχει στον τομέα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Ο κ. Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η πρόταση που μας καταθέτουν οι δύο συνεισηγητές είναι βελτιωμένη σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, αλλά απέχει από αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και ένα σφαιρικό επενδυτικό πρόγραμμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι και στον αέρα, γιατί ακόμη δεν έχουμε το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς στο Συμβούλιο υπάρχουν πιέσεις για να περικοπούν τα κονδύλια που προτείνει η Κομισιόν και όχι να αυξηθούν όπως ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ω κοιόδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας της Αριστεράς συνέβαλα με τροπολογίες μας στο να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν με μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερη γεωγραφική κάλυψη ουσιαστικότερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ισχυρότερο ρόλο στις αναπτυξιακές τράπεζες και περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μέσω των επενδύσεων. πιστεύω όμως ότι συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη για ακόμη πιο φιλόδοξες προτάσεις. γι' αυτό και στην ψηφοφορία θα καταθέσουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σολέ, εκ μέρους των Πρασίνων, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Το InvestEU για μα θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να είναι ένα μέσο για την επίτευξη ε, τη προόδου προ μια βιώσιμη οικονομία. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε την αύξηση των κλιματικών δαπανών, των σχετικών στόχων δηλαδή για βιώσιμε υποδομέ και ε, την. Ε, λήψη των κλιματικών ε, κριτηρίων. Γιατί πρέπει να πετύχουμε του βιώσιμου στόχου ανάπτυξη και του στόχου ε, των Παρισίων. Το InvestEU ελπίζουμε ότι θα τηρήσει την αρχή τη βιώσιμη επένδυση. Και έχοντα αυτά κατά νου, ε, πρέπει να πω ότι δείξαμε ότι οι πυρηνικέ υποδομέ, υποδομέ σε φυσικό αέριο δεν μπορούν να θεωρούνται βιώσιμε. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να εξευρεθεί πολιτική βούληση ώστε ο χρηματοπιστωτικό τομέα να ενθαρρυνθεί να χρηματοδοτεί έργα τα οποία είναι σημαντικά για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Επίσης, είμαστε κάθετα αντίθετοι στη χρηματοδότηση αμυντικών ε, προγραμμάτων με το InvestEU. Υπάρχουν πολύ πιο πιεστικές ε, ε, ανάγκες, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, για τις οποίες απαιτείται η δέουσα προσοχή. Επανέρχομαι στα θετικά και χαιρετίζω την έντονη συμμετοχή των τοπικών περιφερειακών τραπεζών πρόθεσης, που είναι ένας παράγον κλειδί για την ε, επιλογή ε, των σωστών έργων, επειδή γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται επί τόπου, ποιες είναι οι ανάγκες ε, και τέλος ευχαριστώ και τους συνεισηγητές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εξ του FDD ο κύριος Άρνοντ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, θα συμμετέχω εκ νέου στις εκλογές. Το 2014 εξελέγην ε, με μια εντολή τότε για το Brexit και έκτοτε συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθώ πραγματικά να προωθήσω τη βασική αυτή εντολή. Ζητήθηκε ένα δημοψήφισμα για το Brexit. Το δημοψήφισμα για το 2016 ενέκρινε το Brexit αυτό και αυτό ε, εγκρίθηκε από τις μετέπειτα εκλογές. Για τέσσερις φορές λοιπόν οι Βρετανοί πολίτες έχουν επιβεβαιώσει τη βούλησή τους. Για τρία χρόνια λοιπόν τώρα συζητάμε το πρόγραμμα αυτό InvestEU. 40 δισεκατομμύρια από τους φόρους των πολιτών και άλλα 400 δισεκατομμύρια από την, για την τεχνική πλευρά του προγράμματος. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε αν το Ενωμένο Βασίλειο τελικά θα είναι μέλος του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2027 δηλαδή. Δεν μπορεί να το εγγυηθούμε αυτό. Μάρτιος 2019, Ιούνιος 2013, 21 Οκτωβρίου, είχαμε όλες αυτές τις ημερομηνίες ορόσημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ακούσουμε τη βούληση του Βρετανικού λαού που τέσσερις φορές έχουν πει ότι θέλουν να αποχωρήσουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ακριβώς θα ακούσουμε πάλι στις 23 Μαΐου. Και ας ε, θυμηθούμε λίγο και τον Φρανκ ε, Σινάτρα που λέει «Φτάνει σιγά σιγά το τέλος καθώς πέφτει η αυλαία». Καθώς πέφτει λοιπόν η αυλαία θα πρέπει να πούμε ότι δεν καταφέραμε να κινηθούμε με τον δικό μας τρόπο, με τον τρόπο που θέλαμε, αλλά με τον τρόπο που θέλανε οι εκλογείς μας. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κάνουν οι πολιτικοί. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μάλετιτς, τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον κύριο Φερνάντεθ και τον κύριο Γκουτιέρες για την επίτευξη ικανοποιητική συμφωνία όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του προγράμματος InvestEU. Όπως είπε και η παρέχουμε ένα κίνητρο ενθάρρυνση στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με το επόμενο κοινοβούλιο. Έχουμε ξαναμιλήσει για το πρόγραμμα αυτό, γιατί όντως πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία όμως θα έχει η μελλοντική εφαρμογή στα κρατημέλη. Θα πετύχει όταν γίνει πιο ορατό, όταν κατορθώσει να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εμπορικές τράπεζες ή από το Ταμείο Συνοχής. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κοινοτομία, στις νοφείς επιχειρήσεις, Πρέπει να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν σε μέγεθος. Πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι οποίοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας επενδύσουμε λοιπόν σε έργα τα οποία έχουν μια δυναμική, τα οποία μας δεν εκτιμά η αγορά. Χρειάζεται επίσης προσοχή στην γεωγραφική κατανομή των πόρων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αφορούσε κυρίω τι πιο ανεπτυγμένε χώρε. Ήρθε η ώρα όμω να βοηθήσουμε και τι άλλε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Περέση, παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έγκριση του κειμένου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προκρίθηκε με το σχέδιο Juncker και, την, πίεση των σοσιαλιστών. Είναι μερική η νίκη μας εν ώψη της περίοδου 21-27 ε, αλλά χαιρόμαστε έστω και γι' αυτό. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, σίγουρα έχουμε πετύχει μια καλύτερη ισορροπία, διότι υπάρχει μια διευθύνουσα επιτροπή, μια επιτροπή διακυβέρνησης, όπου συμμετέχει και η Κομισιόν και άλλοι θεσμικοί εταίροι, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις κλειδί με οικολογικό επίσης σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγκαλιάσει το θέμα των αηφορικών υποδομών, των επενδύσεων στην κοινωνία και στις δεξιότητες καθώς και στον τομέα του πολιτισμού. Προσοχή όμως, το θέμα της καλύτερης στοχοθεσίας. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των δεσμευσεών μας πρέπει το 40% των επενδύσεών μα να πάει προς το πρασίνισμα της οικονομίας. Και να θυμηθούμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλη μια φορά της δίνει προεξέχοντα ρόλο. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για καλή απόφαση όσον αφορά ε, τα δικαιώματα που θα έχει στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέτς, παρακαλώ. Πρόεδρε, EU αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά κάποιες ενστάσεις που έχω και στις οποίες θα αναφερθώ στο τέλος. Το θέμα είναι λοιπόν να εγγυηθούμε τον στόχο της αντιμετώπιση της μεταφορή του κλίματος. Το θέμα είναι καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Λήψη υπόψη της ανάγκης προστασίας του κλίματος Τώρα, ως προς τις ενστάσεις μου, βλέπω ότι εντάσσεται το πρόγραμμα μας και η άμυνα, καθώς και άλλα έργα τα οποία δεν έχουν σχέση με την προστασία του κλίματος. Βλέπω αεροδρόμια, βλέπω επενδύσεις στην ενέργεια μέσω των ρηκτών καυσίμων. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον του πλανήτη ή όχι. Όταν έρθει ο Μάιο, λοιπόν και η ώρα των εκλογών, σκεφτείτε τι ανάγκε του πλανήτη. Πρόεδρος. Ε, ο κύριο Πασπισίλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συναδελφοί μου ε, με κάλυψαν ήδη λέγοντα πολλά σημαντικά πράγματα όσον αφορά το πρόγραμμα Invest in You, το οποίο προφανώ υποστηρίζω. Θεωρώ ότι το παιδιτικό αυτό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Η εμπειρία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει δείξει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απόλυτα λογικές, σκόπιμες και ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μέσω επενδύσεων σε τομείς οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται αρκετά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το πρόγραμμα Invest in Youth επικεντρωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Χαίρομαι πολύ που θα προωθήσει τους στόχους αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, θα προωθήσει τους περιβαλλοντικούς στόχους και την πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύω ότι στο μέλλον το πρόγραμμα InvestEU θα προωθήσει εν γέννη την ευρωπαϊκή οικονομία, ακριβώς επειδή έχει ένα, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παρέχει εγγύησεις για ιδιωτικά δάνεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω λοιπόν το διάδοχο πλέον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θεωρώ ότι έχουμε αντλήσει πολύ θετικά διδάγματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021 2027. Ευελπιστώ λοιπόν ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό ώστε να αρχίσει να υλοποιείται από το 2020 και μετά. Κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πριν πέντε χρόνια οι σοσιαλιστές όταν κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές απαιτούσαμε το τέλος ε, της λιτότητας ε, των πολιτικών προσαρμογής ε, και ζητούσαμε να δοθεί μεγαλύτερη τόνωση και όθηση στις επενδύσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Φυσικά και ευχαριστούμε και την Κομισιόν και όλες τις πολιτικές ομάδες που προώθησαν το σχέδιο Juncker γιατί αυτό ήταν σημαντικό για να αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια η κρίση. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το βήμα που γίνεται τώρα για τη δημιουργία ενός μόνιμου εργαλείου. Το νέο αυτό Invest Europe, EU, που θέλει να συνεχίσει να τονώνει τι επενδύσει ε, και να τη στηρίζει μόνιμα στην Ένωση, είναι κάτι πολύ απαραίτητο αυτή τη στιγμή που βιώνουμε μια μεγάλη περίοδο στασιμότητας και τελμάτωσης. Ε, το σχέδιο Γιούνκερ, ε, όμως ε, εξακολουθεί να χρειάζεται αντικυκλική πολιτική, όπως αυτή που μπορεί να προσφέρουν αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητέ. Το πρόγραμμα InvestEU είναι μία από τις ε, πιο κεντρικές πλέον πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε θέση να κινητοποιήσει εγγυημένε ιδιωτικές επενδύσεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πολύ πιο φιλικό προβλέψιμο κλίμα για τους επενδυτές. Και βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο μέσω των επενδύσεων αυτών συμβάλλουμε στην ε, ευημερία των πολιτών μέσω καλύτερης οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης, μέσω της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και μέσω της υπεύθυνη χρήσης των πόρων. Επί του παρόντος, οι επενδύσεις βλέπουμε ότι επικεντρώνονται σε ορισμένα μόνο κράτη-μέλη. Συνεπώς, Μέσω του προγράμματος αυτό InvestEU και μέσω των επιλέξιμων προγραμμάτων θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε την κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία προκειμένου να μην αυξάνονται περισσότερο ανισότητε μεταξύ των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, α μην στο ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνήθω αντιμετωπίζουν πολύπλοκε διαδικασίε όταν, όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν επενδύσει. Έρχεται λοιπόν τώρα το πρόγραμμα Invest in EU για να απλουστεύσει τι διαδικασίε αυτέ και να μειώσει τη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να καταφέρουμε να προσελκύσουμε επενδύσει ιδίω σε κάποια μικρά τοπικά προγράμματα, ακριβώ εκεί που μπορεί να επιτευχθεί μόχλευση και εκεί πέρα που μπορούν να συμμετέχουν πολλά κλάστερ ε, επενδυτών. Οι δημόσιε όμως αρχές θα πρέπει και πάλι να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει απαραίτητη δανειοδότηση και το απαραίτητο θετικό ε, κλίμα προκειμένου να προσελκυθούν περισσότερε επενδύσει. Κύριος Ρούμπιχ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κάρας ε, της, ε, του Intergroup για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ο οποίος στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική στρατηγική απόφαση, γιατί θέλουμε να πετύχουμε την ευημερία τους πολίτες και μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ και 25 χρόνια ξέρω πολύ καλά τι ε, έχουν πετύχει τα ΔΕΛΤΑΠΗ ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 500 ε, δις διατέθηκαν και από το 2007 στο 2013 που προωθήσαμε το πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με 2 δις. Και βέβαια έχουμε και το Micro ΜΜΕ 3 δις και το ΕΦΣΙ με 500 περίπου του ε, μαζί με τη μόχλευση. Έτσι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουμε ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 25% τώρα ε, προβλέπεται για επενδύσεις στον τομέα του κλίματος ε. και βλέπουμε ότι έχει κάνει έτσι μία στροφή προοδευτική η Ευρωπαϊκή Όνωση για να ε, είμαστε πρωταγωνιστές ε, και θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μπιενκόφσκα γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο ε, να στηρίξει κανείς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δείξαμε όμως ότι αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστώ και καλή τύχη. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία προσέλκυση προσοχή ε, του Προέδρου Κάτσε Μία, ε, ένα μάλλον έχει τη ο κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα InvestEU πράγματι θα μπορούσε να αποδώσει και θα μπορούσε να συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να στηρίξει την κατάρτιση, να στηρίξει τις δεξιότητες αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν με το σχέδιο juncker διότι η εμπειρία από το ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων ιδίως για την ελλάδα απέδειξε ότι τον πακτολό των χρημάτων τον πήραν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες στην πράξη χρηματοδοτήθηκαν για να αρπάξουν τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. κλασική περίπτωση η fraport η οποία υποτίθεται ότι θα έκανε επενδύσεις στο πλαίσιο μιας δίθεν αποκρατικοποίησης που επέβαλε η τρόικα και έχουμε μια κρατική γερμανική εταιρεία η οποία παίρνει δάνειο 280 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα τόσα από Ελληνική Τράπεζα και αρπάζει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τέτοιου είδους επενδύσεις δεν νομίζω ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Απλά χρηματοδοτούνται οι δίθεν ιδιωτικοποιήσεις άρα λοιπόν το πρόγραμμα πρέπει να πάει σε μια κατεύθυνση στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αυξημένη προστιθέμενη τοπική αξία. ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπιενκόφσκα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, καθώς και για τα θετικά σας σχόλια για το πρόγραμμα και το βασικό συμπέρασμα το οποίο συνάγω από αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει συντριπτική υποστήριξη ε, υπέρ του προγράμματος Investigiu. Πάντως σημειώνω βέβαια και τις πολύ ψηλές προσδοκίες σας και τις συστάσεις σας ε, για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος και θέλω να σας πω ότι θα τις μεταφέρω και θα τις λάβουμε υπόψη αυτές τις συστάσεις ε, κατά την προπαρασκευή του προγράμματος. Ξανά να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές αλλά και όλους όσοι λάβατε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ και για να ολοκληρώσουμε θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή κύριο Φερνάντες. Οι δημόσιες επενδύσει ε, είναι πάρα πολύ σημαντικέ. οι ιδιωτικέ επενδύσει, εξίσου σημαντικέ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, ε, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφύης επιχειρήσεις, να ενισχύσουμε την ε, παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα αμείβονται καλύτερα, με καλύτερους μισθούς, οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες επενδύσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις ε, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Δυστυχώ στη χώρα με την Πορτογαλία. Με το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση και ιδίω ο Πέδρο Μάρκε, ε, ο αρμόδιο υπουργό, δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ ε, για επενδύσει. Το έργο, το σχέδιο Juncker και το InvestEU θα πρέπει να αξιοποιηθούν για δημόσιες επενδύσεις μεταξύ άλλων, όχι μόνο για ιδιωτικέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να βάλουν το λιθαράκι τους. Ε, στο κοινοβούλιο αυτό εγκρίναμε αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για 700 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κινητοποιούνται πάρα πολύ καλή γεωγραφική κατανομή. Έτσι ε, ενισχύουμε και αυτή την πλατφόρμα, αυτό το συμβουλευτικό κόμβο του InvestEU. Πρέπει να υπάρχουν όμως σε εθνικό επίπεδο τέτοιοι κόμβοι που θα βοηθούν τους επενδυτές. Θα μπορούσαν να είναι και περιφερειακές βέβαια οι πλατφόρμες αυτές ε, με στόχο να βοηθήσουμε να διαρθρωθούν τέτοιου είδους επενδυτικές πλατφόρμες και να ε, κατατίθενται καλές υποψηφιότητες για την αξιοποίηση του InvestEU. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε περισσότερη ε, σε επενδύσεις, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Θα πετύχει δηλαδή ε, τους στόχους του αυτό το πρόγραμμα του Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε στο πέρας της θέλω να ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία. Οι ψηφοφορίες θα λάβουν χώρα αύριο. Θα είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση. Ξεκινούμε στις 8 και μισή έως τις 2. Η μέση διάταξη είναι ήδη δημοσιευμένη στον ιστοτοπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω τον κύριο Ρουμπίχ όμως που θέλει τον λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, των ε, βουλευτών που είναι παρόντες θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί προεδρεύατε υποδεγματικά πάντοτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και ελπίζω και υπό άλλες συνθήκες να ξανασυναντηθούμε κατηδίαν ίσω και να έχουμε και άλλες τέτοιες συζητήσεις στην ωραία σας τη χώρα. Ευχαριστώ και πάλι ο Πρόεδρος και κλείνει η συνεδρίαση εδώ σε αυτό το σημείο.